να μην φέρει αντίρρηση στα εφαρμοστικά μέτρα που ανακοινώθηκαν στη χθεσινή έναρξη της Συνόδου. Δεν έχουν υπάρξει αντιρρήσεις, οπότε η σύσταση θεωρείται ότι εγκρίνεται σύμφωνα με τον κανονισμό 105 παράγραφος 6 και θα δημοσιευθεί το, το υιοθετημένο κείμενο αύριο.